οδικές διατάξει που ρυθμίζουν το 2009 2014 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόκειται να τεθούν σε ισχύ από 1η Δεκεμβρίου. Έχουμε 17 έδρες επιπλέον. Και υπάρχει ο 18ος ο οποίος είναι 17 καινούργια μέλη μάλλον είναι ο πρόεδρος και έχουμε έναν 18ο από τις κάτω χώρες που θα 17 καινούριου ε, συναδέλφου διορθώνει τώρα. Οπότε θα σα διαβάσω τα ονόματα και παρακαλώ οι νέοι συνάδελφοι να εγερθούν. Βρίσκονται εδώ στο ημικύκλιο και να του καλωσορίσουμε. ορίσουμε. Φίλοι, νέοι ευρωβουλευτέ, εγερθείτε. Από τη Βουλγαρία, Σβετόσλαβ, Χρήστοφ Μαλίνοφ από την Ισπανία, Βιθέντε, Μιγέλ, Γκαρθέ, Ραμόν. Από την Ισπανία επίση, επαναλαμβάνει Μιγγέλ Γκάρτες Λαμόνι, Ντολόρες Γκαρθία Γιέρο Καραβάγιο, Εύα Ορτίθ Βιγέλα, Σαλβαδόρ Σεδό ή Αλαμπάρτ. Αυτά ήταν τα, οι τέσσερι ευρωβουλευτέ από την Ισπανία, από την Γαλλία δύο ευρωβουλευτέ. Ιβ Κοσέ. Και Ζων Ροατά. Από την Ιταλία, ο Τζίνο Τρεματέρα. Από την Λετωνία, Κάρλις Σαντούρσκης. Από τη Μάλτα, Γιώζεφ Κουσκέρι. Από την Αυστρία, Έβαλτ Στάντλερ και Γιώζεφ Βάντεν Χόλτσερ. Από την Πολωνία, Αρκάντιος Τόμας Μπρατκόφσκι. Σλοβενία, Ζοφία Κουκόβιτς. Από τη Σουηδία, Αμαλία, Anders Dotter, Jens Nilsson. From, from the United... Και από το Ηνωμένο Βασίλειο, McIntyre. Γιάνθια McIntyre. Thank you very much, colleagues. Welcome to the European Parliament, to our hard work. Σας ευχαριστούμε και καλή και σκληρή δουλειά σας εύχομαι. Συνεχίζει ο πρόεδρο. Κύριε. Το επόμενο θέμα το οποίο αφορά πάλι την ενημερωσή σα, το Συμβούλιο δυνάμει τη Διαδόξη 142 μου είπαν σήμερα την κατεπίγουσα διαδικασία όσον αφορά το σχέδιο αποφάσεω το οποίο θα πρέπει να